przewodniczący! Dzień dobry. Paniom i panom posłom. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο, κύριο Μπαρνιέ, Άρχεται η συνεδρίαση. Πρώτο σημείο, δήλωση της Επιτροπής για την ολοκλήρωση